Ε, διάταξη, αγαπητοί συνάδελφοι, το οποίο αφορά δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με οι καζόμενες αποθήσεις στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών στο Φαρμακονήσι που προκάλεσαν ε, θανάτους προσφύγων. Καταρχάς, θα δώσω το λόγο στον κύριο Βενιζέλο. ο οποίο θα προβεί σε δηλώσεις εξ ονόματο του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρίσταμε εδώ ως Προεδρεύων του Συμβουλίου, αλλά φυσικά διατηρώ πάντα την ιδιότητα του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών. Θέλω λοιπόν και υπό τις δύο αυτές ιδιότητες πριν από οτιδήποτε άλλο να εκφράσω την βαθύτατη θλίψη της ελληνικής κυβέρνησης και όλης της ελληνικής κοινωνίας για τις ζωές που χάθηκαν στη θάλασσα στο τραγικό συμβάν στο τραγικό ναυάγιο κοντά στο φαρμακονήσι. έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες πολλά τέτοια δράματα με κορυφαίο το δράμα της λαμπεντούζα. ήδη σήμερα βλέπουμε ειδησιογραφικά να υπάρχει νέα πολύ μεγάλη πίεση στην θαλάσσια περιοχή της λαμπεντούζα παρά τις συνεχείς και άοκνες προσπάθειες που καταβάλουν οι ελληνικές αρχές και ιδίως η ακτοφυλακή υπάρχουν προβλήματα γιατί όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στην προηγούμενη συζήτησή μας για τις πιέσεις που ασκούνται στην βουλγαρία στα χερσαία σύνορα της βουλγαρίας η ελλάδα όπως και οι άλλες νοτιοανατολικοευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες έχει τόσο εκτεταμένες ακτογραμμές έχει να προστατεύσει και να διαφυλάξει τόσο εκτεταμένα ευρωπαϊκά σύνορα ώστε φυσικά δεν επαρκεί πάντα ο μηχανισμός και έχουμε να αντιμετωπίσουμε περιστατικά τα οποία είναι πια τελείως διαφορετικά σε σχέση με αυτά που είχαμε ζήσει στο παρελθόν γιατί η κρίση ο εμφύλιος πόλεμος στη συρία το τεράστιο ρεύμα προσφύγων που έχει δημιουργηθεί προκαλεί τεράστιες πιέσεις και κάθε μέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. η τραγωδία στο φαρμακονήσι είναι λοιπόν ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της σοβαρής μεταναστευτικής πίεσης. να σας δώσω μερικούς αριθμούς από τον αύγουστο του 2012 η κατάσταση στο ανατολικό αιγαίο, στο ανατολικό αιγαίο πέλαγος έχει επιβαρυνθεί εντυπωσιακά. Το 2008 είχαμε 15.000 περιστατικά τα οποία είχαν μειωθεί εντυπωσιακά πριν από την τελευταία έκρηξη στη συρία και το 2011 είχαμε μειωμένα περιστατικά και το. 2012. από τον αύγουστο όμως του 2012 έχουμε μια επιδείνωση. καλύπτει το ελληνικό λιμενικό σώμα η ελληνική εκτροφυλακη μια περιοχή μεγαλύτερη των 2.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη θαλάσσια περιοχή του ανατολικού αιγαίου και η περιοχή αυτή βέβαια περιλαμβάνει ε, μεγάλο αριθμό νησιών και βραχονησίδων. Μέχρι στιγμής έχει προβεί σε ενέργειες διάσωσης 3.120 ατόμων. Αυτό αναλογεί στο 29% όλων εκείνων που έχουν διέλθει χωρίς έγγραφα και χωρίς νόμιμες διαδικασίες τα σύνορα. Στην προκειμένη περίπτωση το τουρκικό αλλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε από τις επίγειες δυνάμεις που εδρεύουν στο φαρμακονήσι ενημερώθηκε αμέσως το περιπλέον σκάφος του λιμενικού σώματος που έσπευσε στην περιοχή υπήρχαν εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες και φτάσαμε σε ένα δράμα πραγματικά γιατί τελικά είχαμε ένα σημαντικό αριθμό ζωών, ανθρώπινων ζωών που χάθηκαν. Το περιστατικό αυτό μας έχει ευαισθητοποιήσει ιδιαίτερα όπως ε, είχε την ευκαιρία να τονίσει ο έλληνας υπουργός ναυτιλίας ο κ. βαρβιτσιώτης σε επιστολή του προς τον επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συμβουλίου της ευρώπης αλλά και προς την κυρία Μάλστρομ, έχει ήδη διαταχθεί και διεξάγεται ανεξάρτητη δικαστική έρευνα για τα περιστατικά αυτά. θέλουμε να διερευνήσουμε πλήρως τα γεγονότα θέλουμε να μάθουμε απολύτως την αλήθεια θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα που να περιορίζει το εύρος και το βάθος της έρευνας αυτής. θα εφαρμοστεί ο νόμος θέλουμε να λειτουργήσει παιδαγωγικά και παραδειγματικά το συμβάν αυτό δεν μπορώ να προδικάσω την έρευνα ξέρω ότι και η frontex όπως έχω διαβάσει στον τύπο έχει τα δικά της στοιχεία και τις δικές της καταγραφές το λιμενικό σώμα έχει παρουσιάσει τα στοιχεία όπως έχουν καταγραφεί ε, μέσα από τους δικούς του μηχανισμούς. σημασία έχει να αντλήσουμε συμπεράσματα από αυτήν την εμπειρία. όπως είχα την ευκαιρία να πω και στην προηγούμενη συζήτηση για την βουλγαρία πρέπει να φανεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της δίκαιης και αναλογικής κατανομής των βαρών πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πίεση η οποία είναι καθημερινή και ταυτόχρονα να διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που είχα την ευκαιρία στην προηγούμενη συζήτηση να παρουσιάσω αρκετά αναλυτικά. είναι μια προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας του εξαμήνου αυτού αλλά και μια προτεραιότητα της ιταλικής προεδρίας του επόμενου εξαμήνου η μεταναστευτική πολιτική η διαμόρφωση μιας ακόμη πιο ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σας θυμίζω ότι ήδη το ευρωπαϊκό συμβούλιο έχει αφιερώσει δύο μεγάλες συζητήσεις τον περασμένο οκτώβριο και τον περασμένο δεκέμβριο η σύνοδος η άτυπη σύνοδος των υπουργών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων πριν από λίγες μέρες στις 24 Ιανουαρίου στην Αθήνα έδωσε την ευκαιρία στους υπουργούς και στην αρμόδια επίτροπο την κυρία Μάλστρομ να συζητήσουν για το τι πρέπει να γίνει και στην μετά την Στοχόλμη εποχή και στόχος μας είναι μέσα και από τις προτάσεις που θα παρουσιάσει η επιτροπή να ολοκληρώσουμε τον ιούνιο στο ευρωπαϊκό συμβούλιο αυτό το σχέδιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. αυτό το επίπεδο του μεσομακροπρόθεσμου προγραμματισμού δεν δίνει βέβαια απάντηση στις καθημερινές πιέσεις τα δράματα την αγωνία την εκμετάλλευση το οργανωμένο έγκλημα που πολλές φορές κρύβεται πίσω από αθώους ανθρώπους από πρόσφυγες που αναζητούν μια καλύτερη τύχη αναζητούν προστασία από τις απάνθρωπες συνθήκες που υπάρχουν στη συρία αλλά και άλλες περιοχές της ε, Μέσα ανατολής και της βόρειας αφρικής. θέλω λοιπόν και εκ μέρους του συμβουλίου και εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης να σας διαβεβαιώσω ότι η έρευνα θα είναι πλήρης η ευαισθησία μας είναι απόλυτη και η συνεργασία με την επιτροπή επίσης ανοιχτή και θέλω να ελπίζω αποτελεσματική. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βενιζέλε. Τώρα θα ακούσουμε τι έχει να μας πει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αγαπητή φίλη και πάντοτε συνάδελφος Σεσίλια Μάλστρομ. Σεσίλια, έχετε το λόγο. Ε, Κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, και εγώ καταρχήν θα ήθελα βέβαια να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου μετά από αυτό το φρικτό γεγονός το φαρμακονήσι και την απώλεια ανθρώπινων ζώων στους συγγενείς και στους επιζώντες. Ξέρουμε το πρόβλημα των μεταναστών στην Ελλάδα και ανησυχούμε. Εδώ και αρκετό καιρό ερχόμαστε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές, ούτως ώστε να τις βοηθήσουμε, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια πραγματικά λειτουργούσα μεταναστευτική πολιτική με βάση τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες. Έχει σημειωθεί πολύ πρόοδος, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα φυσικά. Και θα συνεχίσουμε να βοηθούμε και να υποστηρίζουμε την Ελλάδα στη διαχείριση της μετανάστευσης, στη διαχείριση των συνόρων και των ετούντων άσυλων ακούστηκαν ε, ισχυρότατοι ισχυρισμοί απόθεση προ την Τουρκία. Ε, και αυτό είναι ανησυχητικό. όπω είπε και ο Υπουργό, είμαστε σε επαφή με τι αρχέ συνεχώ, για να διερευνήσουμε το θέμα αυτών των ισχυρισμών και παρακολουθούμε την κατάσταση επιτόπου και μέσω τη παρουσία τη Frontex στην Ελλάδα. Για αυτό το περιστατικό, από τι πληροφορίε που έχουμε μέχρι στιγμή, από ό,τι φαίνεται, ήταν μια επιχείρηση διάσωση. Δεν ήταν μια επιχείρηση ελέγχου των συνόρων. Ο καιρό ήταν πολύ άσχημο και φυσικά είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε ακριβώ τι συνέβη. Φυσικά η απώλεια ανθρώπινη ζωή είναι πάντα παράδεκτη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Το, το επόμενο πρωί εγώ ήμουν στην Αθήνα μετά από αυτό το γεγονό και μίλησα στον Υπουργό Δένδια, που είναι ο Υπουργό Δημόσια Τάξη και Προστασία, και στον Υπουργό Βαρβιτσιώτη, στον Υπουργό Ναυτιλία και θαλασσίων συνόρων. Εξέφρασα τι ανησυχίε μου και του ζήτησα να κάνουν μια ανεξάρτητη έρευνα. Μου είπαν θα το κάνουν. Του παροτρύναμε να λάβουν την, τα απαραίτητα μέτρα, ούτω ώστε παρόμοια περιστατικά να μην συμβούν στο μέλλον. Φυσικά, δράταμε τη ευκαιρία να υπενθυμίσω τώρα στην Ελλάδα και σε άλλου ότι όταν έχουμε επιχειρήσει ε, ελέγχου των συνόρων, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και να σέβονται την αρχή της μη επαναπρόθεση. Η απόθεση είναι παράνομη. Με βάση το διεθνέ δίκαιο και με βάση τους ευρωπαϊκούς νόμους. Οι ετούντες άσυλο στα σύνορα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση ε, στη διαδικασία ασύλου για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να κάνουν αίτηση ασύλου. Ελπίζουμε λοιπόν να γίνει μια γρήγορη Λεπτομερή και διαφανή έρευνα να χυθεί άπλετο φω το τι συνέβη εκείνη την τραγική νύχτα στο Φαρμακονή. Σα ευχαριστούμε. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Θα ξεκινήσει ο γύρο των ομιλητών, οι οποίοι παρεμβαίνουν εξ ονόματο των κοινοβουλευτικών του ομάδων, με πρώτη την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, εξ ονόματο της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ και τον ε, Υπουργό Προεδρεύοντα και την Επίτροπο για τι εξηγήσει που δόθηκαν. Πράγματι το περιστατικό ήταν περιστατικό διάσωση ε, στι 2 η ώρα τη νύχτα. Ωστόσο, από τη στιγμή που ηγέρθησαν κάποιε αμφιβολίε όλος ο φάκελο έχει μεταφερθεί στι εισαγγελικέ αρχές και θα υπάρξει συγκεκριμένη απάντηση. Όμω, κυρία Επίτροπε, επευκαιρία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η Ελλάδα έχει δεχθεί ένα τεράστιο αριθμό, τον οποίο το βάρος δεν μπορεί να φέρει, και δικαίως βεβαίως πρέπει να φέρει το βάρος των προσφύγων και σωστά μνημονεύσατε το άσυλο υπάρχει όμως το θέμα του εμπορίου των ελπίδων των ανθρώπων που γίνεται από την άλλη πλευρά και υπάρχει ανοιχτό το θέμα για το οποίο υπήρξε συμφωνία αλλά για τα τρία πρώτα χρόνια δεν θα υπάρχουν καθόλου επαναπροωθήσεις της τουρκίας. πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα δεν είναι μόνο μιας χώρας. τα σύνορα στην ουσία είναι κοινά γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και η frontex και από την άλλη πλευρά οι γείτονές μας πρέπει να καταλάβουν ότι καλές σχέσεις με την ευρώπη σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνεργάζονται στην καταπολέμηση των δικτύων και των τράφικες ανθρωπίνων ψυχών που θησαυρίζουν στις πλάτες ανθρώπων που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και νομίζω και έχετε βεβαίως την ευθύνη να εισηγηθείτε κυρία επίτροπε και πολύ σωστά έχετε επισημάνει πολλές φορές περισσότερη ευρωπαϊκή προσέγγιση στο ζήτημα αυτό περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών μεγαλύτερη προσπάθεια. η ευρώπη δεν μπορεί να κλείσει τις πόρτες της σίγουρα αλλά δεν μπορεί και να τις ανοίξει διάπλατα υποσχόμενη κακές συνθήκες και γκέτο σε ένα χώρο ειρήνης, ευημερίας και δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γιαννάκου. Τώρα το λόγο εξ ονόματος ε, της ομάδας των έχει για δύο λεπτά η συνάδελφος ε, Μαρία Ελένη Κοπά. Κύριε Πρόεδρε, η τραγωδία με τα 15 θύματα στο Φαρμακονήσι δεν είναι αποκλειστικά ένα ελληνικό πρόβλημα όπω και η τραγωδία με τους 150 νεκρού στη Λαμπεντούζα δεν αποκλειστικά ένα ιταλικό πρόβλημα. Και τα δύο είναι και θα είναι ευρωπαϊκά προβλήματα που αντανακλούν την αδυναμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνει μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική. Η αιμονή στο Δουβλίνο 2 και 3, η άρνηση για δίκαια κατανομή βαρών, με τι παράλληλε απειλέ στι χώρε του νότου για εκδίωξή του από τη ζώνη σέγγεν αν δεν ακολουθήσουν σκληρό και απόλυτο έλεγχο στα σύνορά του οδηγούν σε καθημερινέ ανθρώπινε τραγωδίε με θύματα κυρίω γυναίκε και παιδιά οι οποίε δυστυχώ δεν φαίνεται να λαμβάνουν τέλο. Όμω, κύριε προεδρεύοντα εκείνο που αντίθετα αποτελεί ελληνικό πρόβλημα είναι οι από κάθε πλευρά παράδεκτε και ρατσιστικέ δηλώσει του υπουργού Προστασία του πολίτη νίκου δένδια ότι η χώρα μα έχει την ατυχία να υποδέχεται μετανάστε δεύτερη κατηγορία. παραβλέπει ο υπουργό ότι πρόκειται στην ουσία για ανθρώπου που έρχονται από εμπόλεμε περιοχέ και σε πολλές περιπτώσεις δικαιούνται το καθεστώς πρόσφυγα. δήλωση διπλά απάνθρωπη δεδομένου ότι έρχεται λίγες μέρες μετά τους πνιγμούς στο φαρμακονίσι και χωρίς καν να έχουν αποδοθεί τα σώματα των παιδιών στους γονείς τους. ελληνικό πρόβλημα επίσης είναι οι δηλώσεις του υπουργού ναυτιλίας κ. βαρβιτσιώτη ο οποίος χωρίς ντροπή χωρίς μια συγγνώμη καταγγέλνει τον επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Νιλ μουίζνιεκ ότι θέλει να δημιουργήσει πολιτικά προβλήματα στην ελλάδα και συγχαίρει τον εαυτό του και την υπηρεσία πριν ακόμα ολοκληρωθεί έρευνα. να προσθέσω ακόμα ότι αξιοσημείωτο είναι ότι οι καταθέσει των επιζώντων στην ύπατη αρμοστία του οηε για του πρόσφυγες διαφέρουν παρασάγκα από αυτέ που δόθηκαν στο λιμενικό στην ξηρά. Έγκριτο έλληνα δημοσιογράφος στις 4 δευτέρου αναρωτήθηκε τι είδου κινησμό είναι είναι αυτός; είναι συμπληρώνει η κοινικότητα τη ανεδού και απροκάλυπτης περιφρόνηση του βασικού κανόνα της κοινωνική συμβίωση που δεν είναι άλλος από το σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε Μαρία Ελένη. Έχουμε τώρα παρέμβαση διάρκειας ενός λεπτού από τον συνάδελφο κύριο Χρυσόγελο, εξονόματος των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι χάρηκα που άκουσα τον Προεδρεύοντα και ζήτησε συγγνώμη και εξέφρασε τη λύπη της ελληνικής κοινωνίας γιατί δυστυχώς ενώ συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό μέχρι τώρα δεν είχε ακουστεί μια συγγνώμη. αντίθετα εξεφράστησαν απόψεις για το τι ήταν ακριβώς το περιστατικό πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. χαίρομαι που ανέφερε ο υπουργός ότι εξετάζουμε τι πραγματικά συνέβη και δεν έχει βγει γνωμοδότηση από τα πριν όπως βγήκε ο υπουργός ο άλλος υπουργός ναυτιλίας και είπε περιέγραψε το περιστατικό χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. ελπίζω ότι ο κύριος Υπουργό πράγματι με τις δηλώσεις του ασκεί κριτική στον άλλον υπουργό τον κύριο δένδια ο οποίος μίλησε για ανθρώπους β' κατηγορίας β' διαλογής. αυτό λοιπόν προφανώς πρέπει να αναιρεθεί και ελπίζω ότι ε, εδώ στην ευρωβουλή που πολλές φορές έχουμε μιλήσει για αυτά τα θέματα θα υπάρξει μια άλλη αντίληψη. είναι πράγματι και ευθύνη της ευρώπης όσα συμβαίνουν και αυτό δεν το λέμε μόνο εδώ εμείς μέσα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αλλά το λέει και η έκθεση του συμβουλίου της ευρώπης. δεκαεπτά άνθρωποι πνίγηκαν στη μεσόγειο μέσα σε μια δεκαετία στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην ευρώπη. ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι; είναι κάποιοι άγνωστοι; είναι κάποια παράνομα κυκλώματα; ή πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι οι οποίοι στηβάζονται σε ένα σαπιοκάραβο για να ξεφύγουν από το θάνατο; οι άνθρωποι που πνίγηκαν στην ε, λαμπεντούσα αλλά και σε πολλά άλλα μέρη και στα ελληνικά νερά είναι άνθρωποι που πολλές φορές φεύγουν από εμπόλεμες περιοχές. στο περιστατικό στο Φαρμακονήσι ήταν από το αφγανιστάν και από τη συρία. πρέπει λοιπόν να υπάρξουν διαφορετικές πολιτικές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μην πιέζει η ευρωπαϊκή ένωση για να έχουμε κλειστά σύνορα. πρέπει να υπάρχουν δίωδοι ώστε άνθρωποι που θέλουν να έχουν καθεστώς πρόσφυγα την ασφάλεια να μπορούν να έρθουν νόμιμα να μην πνίγονται. Διακόπτει ο πρόεδρος. Λυπούμε, λοιπόν, υπερβήκατε κατά πολύ τον χρόνο σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, Δυστυχώ ε, είμαι στην πολύ δύσκολη θέση να σας υπενθυμίσω αγαπητοί συνάδελφοι ότι έχουμε πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα ε, και περιορισμένο χρόνο. Εάν ένα συνάδελφο όπω στην τελευταία περίπτωση μιλά διπλάσιο χρόνο από αυτό που, θα του, είχε, που του είχε διατεθεί δεν πρόκειται να ολοκληρώσουμε γέρος. Δεν είναι... αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό του σώματος. Λυπούμε και πραγματικά νιώθω και εγώ αμήχανα, αλλά θα αναγκαστώ να επιβάλλω στον καθένα σας να τηρεί το χρόνο που έχει στη διάθεσή του και αλλιώς ε, αν δεν συμμορφώνονται οι συνάδελφοι μετά από 2-3 δευτερόλεπτα θα αναγκάζομαι να τους κλείνω το μικρόφωνο. Σας ζητώ ε, συγγνώμη κύριε Χουντή γιατί ε, ξέρετε ότι δεν, σας, δεν αναφέρομαι σε εσάς συγκεκριμένα. Εξ ονόματος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ανατολικής Αριστεράς έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Οι πολιτικές και οι πρακτικές κατά μήκο των ελληνικών συνόρων δεν τροπιάζουν μόνο την Ελλάδα, ντροπιάζουν την ευρωπαϊκή ένωση ως σύνολο αυτό γράφει αγαπητοί συνάδελφοι η έκθεση της διεθνούς αμνηστίας τον περασμένο ιούλιο. για το τραγικό γεγονός στο φαρμακονήσι υπάρχουν σοβαρές ευθύνες των ελληνικών αρχών. τέτοιες πρακτικές απόθησης έχουν καταγγελθεί και στο παρελθόν. πρέπει πράγματι να υπάρξει αμερόληπτη έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες. κυρία μάλμστρομ πόσοι άνθρωποι πρέπει ακόμα να χαθούν στη μεσόγειο για να αντιληφθεί η ευρωπαϊκή ένωση ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά την πολιτική τη στο θέμα τη μετανάστευση, στο θέμα του ασύλου στο θέμα τη προστασία θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο το ευρωπαϊκό Έδαφο. πρέπει να υπάρξουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για τη διάθεση των μεταναστών στι ανοιχτέ θάλασσε, να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχή στα σημεία εισόδου και χρειάζεται ένα νέο θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα αριθμίζει πράγματι δίκαια και αναλογικά την πρόσβαση των μεταναστών σε όλες τις χώρες της ευρώπης. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Σα ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Ολοκληρώθηκε ο γύρος των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Περνάμε τώρα στου ε, υπόλοιπου ομιλητέ. Θα δώσω καταρχά το λόγο στην κυρία Χόλμαγερ, η οποία έχει στη διάθεσή τη 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, και πάλι χάθηκαν ζωές ανθρώπων και παιδιών στις ε, ελληνικές ε, οι ελληνικές αρχές μας είπανε ότι ε, μας ενημέρωσαν ότι συμμετείχε και η Frontex και αυτά τα οποία λένε οι ελληνικές αρχές είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που λένε οι ε, πρόσφυγες. Ο, Frontex, ο οργανισμός Frontex ε, δεν μπορεί να κάνει ανάλυση εφόσον δεν είχε συμμετάσχει. Βασίζεται σε αυτά που λένε οι ελληνικές αρχές. Χαιρετίζω λοιπόν τις ε, έρευνες των ελληνικών εισαγγελικών αρχών για να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση. Όσο κάνουν επιχειρήσεις μόνες τους οι εθνικέ ακτοφυλακέ χωρί τη συμμετοχή του Frontex σε τέτοιε καταστάσει, θα έχουμε τέτοια επεισόδια. Γι' αυτό θα πρέπει όλε οι επιχειρήσει να γίνονται από κοινού. Ο Frontex είναι ο ουδέτερο οργανισμό που θα εξυπηρετεί του πάντε. Θέλουμε να σώσουμε του πρόσφυγε, να υποστηρίξουμε τι εθνικέ αρχέ και να εφαρμόσουμε τι ευρωπαϊκέ διατάξει. Επίσης δεν πρέπει να γίνονται εκ των προτέρων ε, ε, κατηγορίες κατά των Ελλήνων ε, δημοσίων υπαλλήλων. Και είναι επίσης απαράκτηση οι κατηγορίες, ε, οι αστοιχείωτες κατά του Frontex. Είναι σαφές ότι υπάρχουν διάφορα κυκλώματα και είναι σαφής και ο ρόλος των τουρκικών αρχών. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, τα κυκλώματα αυτά σε, όλη την, σε όλο το μήκος των συνόρων με την Τουρκία. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφε. Ο κύριος Αρσένης τώρα για ένα λεπτό. Σήμερα νιώθω υποχρέωση δώσουμε τη φωνή μου φωνή στα θύματα της τραγωδίας του Φαρμακονής. Στον Αμπτούλ Σαμπούρα Ζίζη, τον Φαντά Μοχάμετ Αχμάντη, στον Εξάντα Σούφη, για σωθέντες του ναυαγίου που χάσαν όμως τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Λένε, οι λιμενικοί δεν ήρθαν να μας σώσουν, ήθελαν να μας πνίξουν σηκώσαμε ένα μωρό για να το δούνε να δουν ότι έχουμε γυναίκες και παιδιά. οι γυναίκες φώναζαν βοήθεια και οι λιμενικοί τις βρίζανε. θα μας άφηναν να πνιγούμε αν δεν πάθαινε το σκάφος του λιμενικού βλάβη. Ένα σύρο που είχε καταφέρει να ανέβει στο σκάφος του λιμενικού πέταξε ένα ξύλο να πιαστεί ένα παιδί αλλά ο λιμενικός το κλώτσισε. μας έβαλαν να υπογράψουμε χωρίς γερμηνέα καταγγέλλω την υποκρισία την ηθική αυτουργία και τη συνυπευθυνότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που στηρίζουν ακόμα το δουβλίνο ii και που δεν δέχονται να μοιράζονται οι πρόσφυγες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Όμω, οι πολιτικέ εντολέ που δίνονται στου άντρε του ελληνικού λιμενικού να επαναπροωθούνται άτυπα με κάθε μέσο οι πρόσφυγέ πίσω στην τουρκία του μετατρέπει σε δίμιους. και γι' αυτό κύριε βενιζέλο έχετε πολιτική ευθύνη. Σε ευχαριστώ Κρήτονα. Το λόγο για ένα λεπτό έχει ο συνάδελφος Αγκουράκης. Ευχαριστώ. Η τραγωδία στο Φαρμακονήσι είναι αποτέλεσμα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ της έντασης της καταστολής στα σύνορα της ενίσχυσης των δυνάμεων του Frontex. Οι κοινέ επιχειρήσεις καταστολής το μόνο που κάνουν είναι να πολλαπλασιάζουν τα αθώα θύματα είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουν το κύμα μεταναστών γιατί αποτελούν την άλλη όψη της εγκληματικής πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης και των κυβερνήσεων που με τις συμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ευρωπαϊκής ένωσης του νατο και των ηπα ξεριζώνουν ε, εξαθλιωμένους ανθρώπους. σήμερα είναι επίγουσα ανάγκη να σταματήσουν τα νέα μέτρα και η κατασταλτική δράση των μηχανισμών της ευρωπαϊκής ένωσης frontex του ευρωπαϊκού συστήματο επιτήρηση των συνόρων να δοθεί άσυλο ή προσωρινό ανθρωπιστικό καθεστώ σε όσου προέρχονται από χώρε υπεριαλιστική κατοχή ή εμφυλίων πολέμων να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα για όσου θέλουν να πάνε σε άλλο κράτο μέλο τη ευρωπαϊκή ένωση να καταργηθεί ο κανονισμό δουβλίνο 2. τέλο να σταματήσει αμέσω κάθε συμμετοχή τη ελλάδα στι υπεριαλιστικέ επεμβάσει τη ευρωπαϊκή ένωση και του νάτο σε τρίτε χώρε. Σας ευχαριστώ συνάδελφε για ένα λεπτό και τελευταίο σε αυτό το γύρο ο μιλητής ο κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το συμβάν στο Φανακονής ήταν ένα δραματικό γεγονός, μια τραγική στιγμή. Η αντιμετώπιση της λαθρέας μετανάστευσης, ειδικά στη θάλασσα, είναι ένας εξόχως δύσκολος αγώνας. Απ' τη μια πλευρά η συντεταγμένη πολιτεία που οφείλει να προστατέψει τα κρατικά σύνορα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο τις διεθνείς συμβάσεις τις πανανθρώπινες και ευρωπαϊκές αξίες την εσωτερική νομοθεσία συγκεκριμένους κανόνες εμπλοκής. από την άλλη τα αδίστακτα οργανωμένα κυκλώματα εγκληματιών μαφίας δουλεμπόρων αλλά και απελπισμένοι άνθρωποι φοβισμένοι που αψηφούν την ίδια τη ζωή τους. δύο θεμελιώδεις παραδοχές νομίζω ότι μας βρίσκουν όλους σύμφωνο σε αυτή την αίθουσα. πρώτον το δικαίωμα στη ζωή είναι το θεμελιώδες ύψιστο ανθρώπινο δικαίωμα. είναι απόλυτο. δεν νοούνται εκπτώσεις δεν υπάρχουν εξαιρέσεις δεύτερη παράδοχη η προστασία και η ασφάλεια των συνόρων είναι η κορυφαία αποστολή και υποχρέωση της πολιτείας και του κράτους. αυτά είναι τα δύο θεμέλια της πολιτικής που εφαρμόζει η ελλάδα στην αντιμετώπιση του φλέγοντος ζητήματος της λαθρέας μετανάστευσης. αυτή την πολιτική ακολουθήσαμε και τη δραματική νύχτα της 20ης Ιανουαρίου. Τώρα η δικαιοσύνη κάνει τη δική της δουλειά. Η Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Η Ευρώπη οφείλει να κάνει και εκείνη το κομμάτι που της αναλογεί. η δίκαιη αναλογική κατανομή είναι η λέξη κλειδί. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ε, δύο συνάδελφοι οι οποίοι θα λάβουν το λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας Catch the Eye προσέλκυσης της Προσεχής ε, του Προέδρου. Κυρία Βελζιά είναι η πρώτη ομιλήτρια και θα της, διακόψω το, θα της πάρω το λόγο μετά από ένα λεπτό ακριβώς. Μαρή Κριστίν, έχεις το λόγο. Το δράμα του φαρμακονισιού προκάλεσε 12 νεκρούς, 9 ε, γυναίκες και 3 παιδιά. Ζητήθηκε να γίνει αυτή η συζήτηση ε, διότι διάφορες ΜΚΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, με βάση τις μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν, αμφισβητούν την συμπεριφορά των λιμενικών της Ελλάδος υπήρξε μια συλλογική επαναπροώθηση προς την Τουρκία και όχι διάσωση. Την ε, στιγμή που η Ελλάδα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η στάση μας φαίνεται απαράδεκτη και νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί ποιος έχει ευθύνη. Εάν το πρόβλημα αυξάνεται από το 2012 είναι ότι μέσα σε 20 χρόνια πάνω από 20.000 ε, ανθρώπους έχουμε νεκρούς στην ε, Μεσόγειο πρέπει να υιοθετηθεί το κείμενο για τη διάσωση στη θάλασσα πριν το τέλος αυτής της θητείας. 45.000 ε, άνθρωποι έφταναν, έφτασαν στις ακτές της Ευρώπης το 2013. Διακόπτει ο πρόεδρος στην ομιλήτρια. Ο κύριος Μέρφη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Βενιζέλη, η κυβέρνησή σας ε, δεν τα κατάφερε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και αυτή, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, αίμα στα χέρια της. Και προστίθενται αυτοί οι νεκροί στις 20.000 άλλους ανθρώπους που έχουν χάσει τις δύο τελευταίες δεκαετίες τη ζωή τους. Παραγματικοί άνθρωποι. Σας δείχνω την φωτογραφία ανθρώπου που έχασε τη γυναίκα του και τρία, λεπτά, και τρία παιδιά του. Ε, μια άλλη φωτογραφία δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε γυναίκα και τέσσερα παιδιά. Χάθηκαν 12 άνθρωποι σε συνθήκες από ό,τι φαίνεται απάνθρωπης βίαιης μεταχείρισης από άνδρες του λιμενικού οι οποίοι επαναπρόθεσαν βίαιως αυτούς τους ανθρώπους ε, ε, μιλάμε για βίαιες απάνθρωπες πολιτικές τις οποίες ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση και οι ευρωπαϊκές αρχές για να κρατούν σε απόσταση τους πρόσφυγες είναι απάνθρωπο, είναι βίαιο και το σύστημα τα χειρότερα στοιχεία του τα βλέπουμε σήμερα στην Ελλάδα και αυτό το σύστημα πρέπει να ανατραπεί. Ε, Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ολοκληρώσαμε τώρα ε, και το γύρο των παρεμβάσεων στο Catch Θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο κυρία Μάλστρομ για να απαντήσει στις διάφορες παρεμβάσεις ονόματος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Γνωρίζουμε την πίεση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Γι' αυτό, όπως σας είπα στην εισαγωγική μου παρέμβαση, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα όσο μπορούμε. Τεχνική βοήθεια, πρακτική βοήθεια, ανθρώπινη πόρη και σημαντική οικονομική βοήθεια, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μετανάστευσης, ασύλου, ελέγχου των συνόρων που να συνάδει με τους διεθνούς κανόν, διεθνείς κανόνες και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Η τραγωδία που συζητάμε σήμερα στο Φαρμακονήσι Πολλοί αναφέρατε και αυτή τη Λαμπεντούζα πριν από λίγους μήνες που ήμουν εκεί, είδα τα φέρετρα. Είναι κάτι το απαράδεκτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τη αξίζει. Και συμβαίνει κάθε μέρα. Σε μικρότερη κλίμακα, ευτυχώ, αλλά συμβαίνει κάτι τέτοιο κάθε μέρα. Όταν μιλάω με επιζώντες από τη Λαμπεντούζα και από αλλού, λένε ότι ξέρουν ότι ο, ο κίνδυνος να πνιγεί στη Μεσόγειο είναι ίσω. Ε, με, ίσως με το 16-17%. Αλλά όμως παίρνουν το ρίσκο γιατί είναι τόσο απελπισμένοι, γιατί μπαίνουν σε αυτά τα σκάφη, γιατί δεν υπάρχουν νόμιμοι τρόποι για να φτάσουν στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να βρούμε τρόπους για αυτούς τους ανθρώπους, ούτως ώστε να φτάνουν ασφαλώς στην Ευρώπη και στις 28 χώρες. Όχι στις 10 μόνο όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά και 28 χώρες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω επανεκατάστασης ε, ο καθένας πρέπει να αναλάβει το βάρος του. Ε, πρέπει να δούμε τους τρόπους που θα προκρίνουμε μετά τη Στοκχόλμη, την περίοδο μετά τη Στοκχόλμη, αλλά πρέπει όλες οι χώρες να λάβουν την ευθύνη από κοινού. Επίση, πρέπει να συνεργαστούμε με τρίτε χώρε. Κάποιο ανέφερε την Τουρκία. Πριν τα Χριστούγεννα ήμουν εκεί και υπέγραψα με τον Τούρκο Υπουργό τη Συμφωνία Επανεισδοχή, που ελπίζουμε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, ε, επεκτείνουμε τη συνεργασία μα σε άλλε χώρε. στην Ισία, Μαρόκο, ε, Αίγυπτος και Λιβύη. Θα έπρεπε, αλλά είναι δύσκολο, λόγω του ότι η κατάσταση είναι όπω την ξέρετε. Δεν είναι εύκολο να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή με αυτέ τι χώρες. Το να ε, καταπολεμήσουμε τα κυκλώματα λαθρεμπόρων και να δημιουργήσουμε αξιόπιστε πολιτικέ ε, μετανάστευση. Επίσης και σε μεγαλύτερη κλίμακα, με την ε, Frontex, σε επιχειρήσει διάσωση Και από την αρχή του 2014 Έχουμε την ε, επιχείρηση Eurosur, όπου προσπαθούμε να δούμε και τα πιο μικρά σκάφη, τις βάρκες και να σώσουμε τους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αλληλεγγύη στην Ευρώπη, αλλά και περισσότερη ευθύνη, διότι αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Η πολιτική μας θα πρέπει να συμμορφώνεται απόλυτα ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, να επιτρέπουμε στους ανθρώπους μας να φτάνουν στα σύνορα για να ζητήσουν άσυλο. Δεν είναι έγκλημα, δεν είναι παράνομο το να ζητάς άσυλο. Το προβλέπει και η Σύμβαση της Γενέβης και προστατεύει τους ανθρώπους αυτούς. Το πολιτικό κλίμα όμω σήμερα δεν είναι πολύ ευίωνο για κάτι τέτοιο. Αν μπορούμε όμως να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους ε, στην περιοχή μας, είμαστε, τα πάμε καλά. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε είναι πρόβλημα. Είναι φρικτή αυτή η θάνατη στην, ε, στο φαρμακονήσι. Οι ισχυρισμοί που βαραίνουν την Ελλάδα είναι πραγματικά ανησυχητική και θέλω ε, να χυθεί το φως μέσω της έρευνας, η οποία θα πρέπει να είναι γρήγορη και ανεξάρτητη, για να, δούμε, για να δούμε τι έγινε αυτή την ε, άσχημη νύχτα. Σας ευχαριστώ Σεσίλια. Θα ολοκληρώσουμε την παρέμβαση εκ μέρου του Συμβουλίου του φίλου μα κυρίου Βενιζέλ. Παρακαλώ κύριε Βενιζέλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να πω κυρίε και κύριοι βουλευτέ ότι στην μακρά κοινοβουλευτική μου θητεία έχω μετάσχει αρκετές φορές δυστυχώς σε συζητήσεις στο εθνικό κοινοβούλιο όπου ζητήματα ζωής και θανάτου ανθρώπινα δράματα γίνονται αντικείμενο μιας πολιτικής συζήτησης με μεγάλη ευκολία. θα μου αναγνωρίσετε σας παρακαλώ πολύ τουλάχιστον την ίδια ευαισθησία με την καθεμιά και τον καθένα από εσά στα θέματα αυτά στο σεβασμό της ανθρώπινης αξίας και στην αυθόρμητη συναισθηματική και ηθική αντίδραση απέναντι σε κάθε πράξη που έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων και ιδίως τον θάνατο μικρών παιδιών. δεν θέλετε να προδικάσει η ελληνική κυβέρνηση το αποτέλεσμα της έρευνας και δεν το προδικάζει δεν πρέπει να το προδικάσει όμως και κανείς άλλος που μετέχει σε μια πολιτική συζήτηση δημοκρατική κοινοβουλευτική. εμπιστευόμαστε την ανεξάρτητη έρευνα και μάλιστα την εισαγγελική δηλαδή την δικαστική έρευνα γιατί στην ελλάδα η εισαγγελία ανήκει στην δικαιοσύνη αποτελείται από ισόβιους ανεξάρτητους δικαστές που δεν έχουν καμία επαφή με την εκτελεστική εξουσία. θα ερευνηθούν όλα τα περιστατικά και θα εφαρμοστεί αυστηρά ο νόμος. επίσης επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι η κυβέρνηση δια του συμβουλίου της ευρωπαϊκής ένωσης εκφράζεται εδώ με αυτά που είχα την τιμή να σας πω εγώ. αυτά που σας είπα υπερκαλύπτουν τις δηλώσεις άλλων συναδέλφων μου που έγιναν τις προηγούμενες μέρες. άλλωστε μετά το δραματικό αυτό περιστατικό στο φαρμακονήσι λίγες μέρες μετά στις 24 Ιανουαρίου η κυρία Μάρστρομ είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί στην Αθήνα και με τον κύριο Δένδια και με τον κύριο Βαρβιτσιώτη τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Ναυτιλίας. Έχει μια πλήρη εικόνα για την άποψή τους. Ναι, δεν μπορούμε πράγματι να κατατάσσουμε σε διαφορετικές κατηγορίες ποιότητας τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους εξητούντες άσυλο δεν μπορούμε να κατατάσσουμε σε κατηγορία κανέναν άνθρωπο. η ανθρώπινη αξία είναι πάντα η ίδια. είναι η βασική αρχή της ισότητας του κάθε ανθρώπου λόγω της φύσης του ως ανθρώπου και αυτό αφορά φυσικά και τους μετανάστες και τους πρόσφυγες όλους μας. ο κύριος βαρβιτσιώτης ανέφερα προηγουμένως ο έλληνας υπουργός ναυτιλίας για όσους δεν ξέρουν ποιος είναι ο κύριος βαρβιτσιώτης έστειλε ήδη επιστολή στον επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συμβουλίου της ευρώπης και του δηλώνει την διαθεσιμότητα απόλυτη συνεργασία των ελληνικών αρχών και με το συμβούλιο της ευρώπης. συναντήθηκα σήμερα το πρωί με τον γενικό γραμματέα του συμβουλίου της ευρώπης και συζητήσαμε με πρακτικό και συγκεκριμένο τρόπο για το πώς μπορεί και πρέπει να οργανωθεί η συζήτηση αυτή η συνεργασία αυτή με απόλυτο σεβασμό στις αρμοδιότητες και τις ευαισθησίες του επιτρόπου η κυρία Μάστρομ έκανε στην αρχή της τοποθέτησής της μια πολύ σημαντική διάκριση διαχώρισε τις επιχειρήσεις ελέγχου συνόρων από τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και χαρακτήρισε το συμβάν στο φαρμακονήσι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που διέπεται από πολύ γνωστούς κανόνες είτε της σύμβασης του σικάγο είτε της σύμβασης του αμβούργου έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ στην ελλάδα με τα ζητήματα έρευνας και διάσωσης και για λόγους ανθρωπιστικούς αλλά και για λόγους σχετιζόμενους με την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. και συμφωνώ απολύτως ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία επαναπροώθηση πλην των προβλεπόμενων σε συμβάσεις επανεισδοχής διαδικασιών. από την άλλη μεριά η αλήθεια είναι ότι αν η ευρωπαϊκή ένωση με την επιτροπή με την frontex δεν παρεύει αποτελεσματικά στα σημεία εκείνα από τα οποία ξεκινάνε τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο με αποτέλεσμα να κερδίζουν πολλά χρήματα οργανωμένες συμμορίες δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. πράγματι το ιδεώδες θα ήταν να μπορούμε να εξετάσουμε αιτήσει παροχής ασύλου στις ακτές από τις οποίες ξεκινούν αυτά τα πλοία που δεν σέβονται τους ανθρώπους που μεταφέρουν και τους εκθέτουν σε δραματικό και θανάσιμο κίνδυνο. πράγματι θα μπορούσαν αποστολές της ευρωπαϊκής ένωσης να εγκατασταθούν στις ακτές της τουρκίας της λιβύης της αιγύπτου και να κάνουν τον έλεγχο αυτό. και πράγματι αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά μηχανισμών αυτούς τους μηχανισμούς πρέπει να τους δούμε να λειτουργούν όχι στα ευρωπαϊκά σύνορα αλλά στα απέναντι σύνορα είτε θαλάσσια είτε χερσαία. αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε για μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Αλλιώ θα είμαστε θύματα της βαθιά ανισότητας που υπάρχει ανάμεσα στι χώρε του νότου τι μεσογειακές χώρε, τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ευρωπαϊκής ένωσης τις χώρες που έχουν χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμών και τις χώρες βέβαια που είναι στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα και δεν έχουν τέτοιες πιέσεις. μιλάμε πάρα πολύ συχνά για αλληλεγγύη μιλάμε πάρα πολύ συχνά για δίκαιη και αναλογική κατανομή των βαρών αλλά οι πιέσεις είναι τελείως διαφορετικές και τελείως άνισες. πιστεύω ότι όλοι εκφραζόμαστε με ειλικρίνεια με ευθύτητα και από την άποψη αυτή η συζήτηση βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ προκειμένου να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. από την άποψη αυτή προφανώς και ο καθένας αναλαμβάνει την πολιτική του ευθύνη και πρέπει να ομολογήσω κι εγώ ότι στη διάρκεια της πολιτικής μου ζωής έχω πολλές πολιτικές ευθύνες ακόμη και για την παρουσία εκλεκτών συναδέλφων στην αίθουσα αυτή. σας ευχαριστώ πολύ. τον κύριο Βενιζέλο με την παρέμβαση του οποίου ολοκληρώνεται η συζήτηση και ερχόμεθα στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης στην κοινή συζήτηση των εκθέσεων προόδου για τα Βαλκάνια και συγκεκριμένα δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την έκθεση προόδου του 2013 για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη